Dear colleagues, let us begin. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε. Καταρχήν με τις ανακοινώσεις σχετικά με τις αποφάσεις που έλαβαν οι συντονιστές χτες. Καταρχήν διορισμός ηγητών. Αποφάσισαν να ορίσουν τον κύριο η εισηγητή για δύο γνωμοδοτήσεις. Πρώτον για την αποφάση Συμβουλίου για την ε, σύναψη ε, συμφωνίας του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη τρομοκρατίας. Και δεύτερον, τα πρόσθετα πρωτόκολλα αυτής της συμφωνίας. Δεύτερον, οι συντονιστές ε, αποφάσισαν να μην γνωμοδοτήσουμε για την ΑΦΚΟ για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και για την ΕΚΟΝ για την ε, αυτόματη υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικά θέματα σχετικά με τις ε, ε, διασυνορικές διευκολύνσεις. Τέτα, τρίτον, αποφασίσαν να γράψουν επιστολή στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου για την Task Force για την επικορικότητα, την αναλογικότητα και κάνοντας λιγότερα πιο αποτελεσματικά. Τέταρτον, αποφάσισαν να καλέσουν τον εκτελεστικό διευθυντή, τον απερχόμενο εκτελεστικό διευθυντή της EU ε, σε μια επόμενη συνεδρίασή μας στο τέλος της θητείας του, περίπου τον Απρίλιο του 2018. Τώρα, συνεχίζουμε με τις πληροφορίε. Ψηφίζουμε καταρχήν για την Έκθεση Βιέφκα, Διεθνή Δικαιοδοσία, Αναγνώριση και Εκτέλεση Αποφάσεων σε γαμικέ Διαφορές. Πρώτη 93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8 και 9 και υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ. 6, ε, 96 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 99. Όχι. Όχι. 100 ε. υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 102 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται Εκατόν τρία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 9 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Πέτη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 515 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 115 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 117 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ελέγχουμε ε, ηλεκτρονική επιβεβαίωση για την 117 We have one too much, no? Yes, we have 25. We should have 25, no? Okay, we close. Λήξη ψηφοφορίας εγκρίνεται. 120 υπέρ. Κατά. Ναι, 120 είναι. 120 ξανά υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 5-16 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 121 υπέρ. Κατά. εποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 139 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 145. Με την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Ας ε, ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. ε, περισσεύει μία κάρτα. Από το ΕΛΚ. Ωραία. Τώρα είναι εντάξει. Τώρα είμαστε εντάξει. Από το ΕΛΚ προερχόταν αυτός ο, ο, ο υπέρμετρος.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 εγκρίνεται 18 υπέρ 7 κατά 145 πάμε στην Yes. Adopted. 146. 146 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πέτη 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 163 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική εξακρίβωση. It has been adopted. Uh, seven εγκρίνεται 17 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 172 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 174 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 175 υπέρ κατά ηλεκτρονική εξακρίβωση. Απορρίπτεται. Εκατόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 177 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 178 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 179 υπέρ κατά ηλεκτρονική εξακρίβωση για την 179 εγκρίνεται 180 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική πρόταση 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 188 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 όχι 189 και 28 της πέτη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 190 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 529 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 51 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά ηλεκτρονική εξακρίβωση για τις 45 It has been rejected. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε μαζί τις 2 και 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική παριθμό 2 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 56 και 57 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά εποχέ, εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά εποχέ, εγκρίνεται. 67 υπέρ. Κατά εποχέ εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά Ας το ελέγξουμε. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Το ελέγχουμε. Εγκρίνεται. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 76 και 11 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 77 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά εποχές το ελέγχουμε 12. Απορρίφθηκε. 80. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 82. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, ας το ελέγξουμε. τη γνώμη δεν θα έπρεπε να την έχουμε ψηφίσει, είναι ασύμβατη με την 80 και την 5 12. Συνεπώς δεν θα έπρεπε να την έχουμε θέσει σε ψηφοφορία την 82. Περνάμε στην 83. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 84. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 85. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5-13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5, 88 και 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τέσσερα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ωραία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά στο σύνολο του κειμένου. One, yes. Close the vote. Κλείνω τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται με Συγχαρητήρια στον κύριο Σβιεύκα. Τώρα ψηφίζουμε επί της έκθεσης του κυρίου Βέλκεν. για τους ε, κανόνες περί ε, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ε, και σε σχέση με τις εκπομπές. Είμαστε στη συμβιστική παριθμόν 1. Υπέρ. Κατά. Παρακαλώ να ελέγξουμε για να είμαστε βέβαιοι. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά. Το ίδιο ήταν, όχι. Αναλέγξουμε λοιπόν ηλεκτρονικά. Μάλιστα, εγκρίθηκε. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα, η ίδια πλειοψηφία, 13 προς 12. So now we are at, uh, yes, Mrs. Μάλιστα, κυρία Στεράς. Εγώ ψήφισα κατά λάθο υπέρ, ενώ ήθελα να ψηφίσω κατά. Επαναλάβατε παρακαλώ, ναι. Ήθελα να ψηφίσω κατά ενώ ψήφισα υπέρ. Α, είναι πολύ αργά τώρα. Λυπούμε. in Είμαστε στην Κουλτ 16. Ο κύριος Λεμπρετό. σε μια προηγούμενη επιτροπή ζουρή, μια από τις απολογίες μου είχε ψηφιστεί, κάποιος ζήτησε να ξαναψηφίσουμε, ξαναψηφίσαμε και απορρίφθηκε. Οπότε με εντυπωσιάζει που σήμερα δεν ισχύει ο ίδιος κανόνας. Πιστεύω πως πολλοί μεταξύ ημών θυμόμαστε τι είχε συμβεί τότε. Είναι σοβαρό το πρόβλημα. Ε, δηλαδή οι κανόνες να μεταβάλλονται ανάλογα με το σε ποια ομάδα ανήκει αυτός το οποίο η, η τροπολογία ψηφίζεται. Let us check. Ας ελέγξουμε. Do You want to check? Compromise two. Let's vote again. Okay. Ας ξαναψηφίσουμε λοιπόν τότε την συμβαστική 2. Εντάξει. Electronically, please. Ηλεκτρονικά παρακαλώ να ψηφίσουμε. Okay. In that case it has been rejected. Απορρίπτεται σε αυτή την περίπτωση λοιπόν. And that means that we continue by... Συνεχίζουμε λοιπόν. Αυτό σημαίνει ότι αφού απορρίφθηκε θα πρέπει να ψηφίσουμε όλες τις τροπολογίες 193, 194, 195 και 192 από κοινού. Υπέρ, κατά, αποχές, πρέπει να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Λείπουν τρεις ψήφοι. Μία ακόμη. Ωραία. Πέρασε τις ε, ψηφοφορίες. Και απορρίφθηκε. 197 υπέρ. Κατά. 197. Είμαστε στην γκρίζα ζώνη. Μετά από τη συμβιβαστική 2 υπάρχει αυτή η γκρίζα ζώνη. 197 λοιπόν. Περκατά. Πολύ λίγα χέρια βλέπω να σηκώνονται. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. It has been rejected. Απορρίφθηκε. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 198 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. One more. Άλλη μία. Απορρίφθηκε. 202 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αυτό ήταν ξεκάθαρο τώρα. 11 υπέρ. Κατά. Αυτό θα το ελέγξουμε. Κατά τη γνώμη μου, απορρίφθηκε. Αλλά να το, να το εξακριβώσουμε. Yes. Rejected 199 in favor. Απορρίφθηκε 199 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 200 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 201 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 203 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 16. Απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά. Έλεγχος ηλεκτρονικός. Κατά τη γνώμη μου απορρίφθηκε, αλλά... Μάλιστα, απορρίφθηκε. Εναλλακτική συμβιβαστική α, υπέρ. Κατά. Φαίνεται να περίφθη, αλλά θα ελέγξουμε να ψηφίσουμε, συνάδελφοι. It was adopted. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε και πάλι. Μάλιστα. πορύφθηκε. Οπότε πάμε. Α, έχουμε εναλλακτική Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εδώ θα ελέγξουμε. Ποια ήταν η γνώμη σου. Απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε. Πάμε στην 223. Α, ναι, ναι, έχετε δίκιο. Απορρίφθηκε, άρα πάμε στην εναλλακτική C. Εναλλακτική C, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Uh, λοιπόν, συνάδελφοι, συγγνώμη, έκανα λάθο. Πρέπει να ψηφίσουμε την γκρίζα ζώνη ανάμεσα σε αυτά που ψηφίσαμε τώρα. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε την 222 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 220 και 19 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 221 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται θέλετε να ελέγξουμε μάλιστα πάμε για να ελέγξουμε τη 221 Απορρίφθηκε όντως. Τώρα πάμε στην 223. Ε, υπέρκατα αποχές απορρίπτεται. Είμαστε στην εναλλακτική συμβιβαστική D. Υπέρ κατά ελέγχουμε παρακαλώ για να είμαστε βέβαιοι.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 Τρεις σελίδες περίπου πιο πέρα. Το βρήκατε όλοι? Όχι. Είναι η 265. Άρθρο 2, παράγραφος 2, α, 2β. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 269 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται εναλλακτική συμβιβαστική ή υπέρ κατά αποχές εκρίνεται Α, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά αφού θέλετε συμβιβαστική ή έλεγχος ηλεκτρονικός Εγκρίθηκε. Τώρα περνάμε στην συμβιβαστική 8. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 304 και 305 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 307 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 310 υπέρ κατά να ελέγξουμε την 310 ηλεκτρονικά παρακαλώ Απερίφθη. Συμβιβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εναλλακτική F υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. εγκρίνεται 318 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 320 μέχρι 35 υπέρ κατά πρέπει να ελέγξω και πάλι εγκρίθηκε 327 έχει αποσυρθεί. Ψηφίζουμε για την 328 και την 28. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 329 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 330 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 331 και 332 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αναλλακτική συμβιβαστική G. Υπέρ κατά. Να ελέγξουμε αυτή παρακαλώ. Εγκρίνεται. Περνάμε στην 32. Ε, Ήτρε 2, συγγνώμη. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 10, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται ήτρε 4 υπέρ τι έκανα λέει τι ξέχασα α ναι με συγχωρείτε ευχαριστώ που με ειδοποίησατε λοιπόν ε, τροπολογία 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται κουλτ 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά να ελεγξουμε 30-32 ηλεκτρονικά παρακαλώ. Απορρίφθηκε. Ήτρε 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αναλλακτική H. Alternative H in favor. Εναλλακτική H υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προχωράμε τώρα στην εναλλακτική συμβιβαστική I. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 53 βρήκατε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβιβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές <coughs> απορρίπτεται. Οπότε πρέπει πάλι όλες αυτές να τις ψηφίσουμε. Μάλιστα. Κουλτ 5 υπέρ. Πρέπει πάλι να περάσουμε όλη την κρίζα ζώνη. Κουλτ 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. is being rejected. Απορρίφθηκε. 58 ε, in favor, 58 ε, μέχρι και 59. 58 και 59 από κοινού υπέρ. Τα κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αναλλακτική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 15 όχι έχει καταπέσει. Πάμε στην εναλλακτική κάπα και υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οπότε προχωράμε στην εναλλακτική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εναλλακτική M υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εγκρίθηκε Πάμε στην εναλλακτική συμβαστική νη υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 111 και 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 112 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται εναλλακτική συμβιβαστική όμικρον ο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά ελέγχουμε την 7 παρακαλώ εγκρίθηκε συμβιβαστική 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Εναλλακτική πι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Είμαστε στη συμβιβαστική 2. 22, συγγνώμη. Υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε. Ξέρω ότι είναι κουραστικό, λέει ο πρόεδρος, αλλά είναι σημαντικό να σηκώνετε τα χέρια σας. Εγκρίνεται. 140 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 141 και κουλ 13 υπέρ κατά αποχές α, απορρίπτονται 142 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 143 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 144 υπέρ απορρίπτεται 145 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 146 και 15 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε. Δεκτές 148 και 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 149 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 152 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτον, απορρίπτεται. Ήταν και άλλες δύο μαζί. 153 μέχρι και 17 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτές. 154 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 155 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. Να ελέγξουμε. Θέλετε να ελέγξουμε. Ωραία. Το 155. Απορρίπτεται. Συγγνώμη. Εναλλακτική συμβαστική R υπέρ κατά να την ελέγξουμε. δεκτή 166 μέχρι και τη 15 υπέρ κατά αποχές δεκτές εναλλακτική συμβαστική S υπέρ κατά αποχές δεκτή 175 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται εκατόν εβδομήντα επτά υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 178 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβαστική 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Εναλλακτική συμβαστική ταφ υπέρ κατά αποχές δεκτή. 189 και 190 υπέρ κατά αποχές δεκτές. Και τώρα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά το τροποποιηθέν σχέδιο έκθεσης άρχεται. Εγκρίνεται. Συγχαίρουμε τον κύριο Βέλκιν και τώρα να ψηφίσουμε επί της αποφάσεως να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. ηλεκτρονικά και εδώ. Ναι, άρχεται η ψηφοφορία βεβαίω. Εγκρίνεται. Λοιπόν, μπορώ να συγχαρώ τον κύριο Βόλκεν. Βεβαίω και το συγχαίρω. Όχι κατά ανάγκη. Yes, the four, the four. One, one after the other. Now we continue our vote. Συνεχίζουμε τη ψηφοφορία. Συνάδελφοι, συνάδελφοι. We continue the... Λοιπόν, έχουμε και άλλες ψηφοφορίες. να ψηφίσουμε την έκθεση Τζαμπάσκι για την απόφαση του Συμβουλίου για να, το, να ε, ε, δοθεί άδεια στο Λουξεμβούργο και τη Ρουμανία. Παρακαλώ ησυχία. Παρακαλώ ησυχία. Σας παρακαλώ όλους ησυχία. Λοιπόν, έκθεση Τζαμπάσκι απόφαση του Συμβουλίου που εξοδοτεί το Λουξεμβούργο και τη Ρουμανία να αποδεχθούν ε, προ το συμφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση την ε, ένταξη τη Γεωργία και τη Νότια Αφρική στην σύμβαση τη Χάη. Υπέρ παρακαλώ. Α, όχι, α, όχι, ηλεκτρονικά, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, λάθο. One more. Λείπει ένας. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στο σημείο 19. Επίση ηλεκτρονικά παρακαλώ. Εγκρίνεται. Σημείο 20. ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται και το σημείο 21 ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται. Τώρα, έχουμε τώρα τη δική μου έκθεση για τον κανονισμό, για την αμοιβαία αναγνώριση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 αποχές απορρίπτεται 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52 υπέρ κατά αποχές δεκτή 53 υπέρ κατά αποχές δεκτή 54 υπέρ κατά αποχές δεκτή 55 υπέρ κατά αποχές δεκτή 56 υπέρ κατά αποχές δεκτή 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59 υπέρ κατά αποχές δεκτή 60 υπέρ κατά αποχές δεκτή 62 υπέρ κατά αποχές δεκτή 64 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές δεκτή 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 65 και 66 από κοινού υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 67 υπέρ κατά αποχές δεκτή, δεκτή να είστε καλά 10 υπέρ κατά Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Ε, ξεχάσαμε τα 68 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή 69 υπέρ κατά αποχές δεκτή 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή 70 υπέρ κατά αποχές δεκτή 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά να ελέγξουμε τη 16 Λείπει ένα, Καλός. Πέρας. Εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε παρακαλώ Λείπει ένας ακόμη. Όχι. Καλώς. Εγκρίνεται. Λειτουργούν σωστά όλα τα μηχανήματα. Γιατί πάντα λείπει ένας. Λοιπόν, 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1 και 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή 32 υπέρ κατά αποχές δεκτή 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή 33 υπέρ κατά αποχές δεκτή 34 υπέρ κατά αποχές δεκτή 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή 36 υπέρ κατά αποχές δεκτή 37 υπέρ κατά αποχές δεκτή 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές δεκτή 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ηλεκτρονικά τώρα ε, το σύνολο της έκθεσης One more maybe. Λείπει πάλι ένας. Όχι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Λοιπόν, να συγχαρώ λοιπόν τον εαυτό μου. <laughs> Ε, one, last vote. Και μία τελευταία ψηφοφορία ηλεκτρονικά για την έκθεση Μαστάλκα. Άρχεται. Εγκρίνεται και να συγχαρούμε και τον κύριο Μαστάλκα. We did it almost. 11. it. And, I love On time. On schedule. yes. So what are we doing now?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 Dear we continue by... Αγαπητοί συνάδελφοι, να περάσουμε στο σημείο 24. Να εξετάσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης για την ισορροπία μεταξύ εργασίας και άλλων καθηκόντων των γονέων και φροντιστών. Η κυρία Μπερζεγό, που είναι η, εισηγήτρια, η συντάκτρια της γνωμοδότησης. Παρακαλώ. Mrs. Ίσως η κυρία Κάουφμαν. Η κυρία Η κυρία Μπεζογό, παρακαλώ, ε, σας έχω δώσει το λόγο. Α, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, φλία ρούσα, είμαι αδιόρθωτη. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η πρόταση οδηγίας ε, ε, προτείνει μια πιο ευρεία προσέγγιση για την ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της κοινωνίας ε, τα τελευταία χρόνια. Η πρόταση αυτή θέλει να αντιμετωπίσει το θέμα της υποεκπροσώπησης των γυναικών στην αγορά εργασίας και να στηρίξει την ε, εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους, ούτως ώστε να μπορούν να συνδυάσουν την οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή. Καθορίζει τα ελάχιστα κριτήρια για να επιτευχθεί η ισορροπία ανδρών γυναικών ε, όσον αφορά τις ευκαιρίες που θα έχουν στην αγορά εργασίας και στο πώς αντιμετωπίζονται στην εργασία όσοι ε, εργάζονται μερικώς είναι κυρίως γυναίκες. 32% είναι γυναίκες, ενώ είναι μόνο 8% οι άνδρες. Και αυτό γιατί είναι δύσκολο να συνδυαστεί η καριέρα με την, ε, με την οικογενειακή ζωή. Και πολλές φορές υπάρχουν και διαφορές στις αμοιβέ και στις συντάξεις. Πολύ μεγάλες διαφορές. Το παρόν νομικό πλαίσιο της Ένωσης και των κρατών μελών δεν προβλέπει αρκετά, ούτω ώστε οι άνδρες να αναλαμβάνουν ισότιμα τις οικογενειακές φροντίδες μαζί με τις γυναίκες. Είναι πήγον να καλύψουμε αυτό το κενό. Η συγκίτριά σα ε, συμφωνεί με τους συγκεκριμένους στόχους τη οδηγίας. Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε τις δυνατότητες πρόσβασης ε, στα μέτρα που θα μας επιτρέψουν αυτή την ισορροπία και για να μπορούν να παίρνουν περισσότερο οι άνδρες οικογενειακή άδεια και πιο ευέλικτες μορφές εργασίας. Το θέμα των ε, αμοιβών είναι ουσιώδες όταν έχει κανείς οικογενειακή άδεια για να μπορούν να υποφελούνται ισότιμα τα δύο φύλλα. Αυτό δεν ισχύει σήμερα γιατί είναι γελίες οι αμοιβέ για τις ε, ε, γονικές άδειες. Και αυτό σημαίνει ότι υπονομεύονται οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί. Η πρόταση της Επιτροπής θεωρεί ότι πρέπει να λαμβάνουν ε, ίδια αμοιβή με το αν ήσαν σε αναρωτική άδεια όσοι λαμβάνουν γονική άδεια. Συμφωνώ λοιπόν και θέλω να πάμε πιο μακριά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υπάρξει ισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών για να μπορούν ισότιμα λοιπόν να λαμβάνουν αυτές τις γονικές άδειες ή τροπολογίες αυτές έχουν κοινή γραμμή να προστατευτούν βεβαίως τα παιδιά πρώτα απ' όλα να υπερισχύει το ε, συμφέρον των παιδιών γιατί σίγουρα ε, το παιδί έχει συμφέρον να ανατραφεί και από τους δύο γονείς εξίσου. Θεωρώ λοιπόν αναγκαίο οι άνδρες και οι γυναίκες να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στην οικογενειακή φροντίδα. Αυτό είναι δυνατό. Εάν ε, δεν υπάρχουν ανισότητες στην εργασία και αν υπάρχει κοινή ευθύνη στην φροντίδα των παιδιών και των άλλων μελών της οικογένειας που χρειάζονται βοήθεια. Ωστόσο, να μην ξεχάσουμε ότι υπάρχουν και περιορισμοί και ανάγκες των εργοδοτών, ιδίω για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις όπου έχουμε δύο ή τρεις εργαζόμενους. Διότι αν λάβει ένας από αυτούς γονική άδεια, μπορεί η επιχείρηση να κινδυνεύσει η επιβίωσή της. Πρέπει, λοιπόν να προστευτούν και οι ε, εργοδότες και να μην υπάρχουν καταχρήσεις. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει ακριβώς να υπάρχουν επαρκή δικαιολογητικά και ε, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν αυτές οι γονικές άδειες στους εννέα μήνες. και θα πρέπει να πλησιωθούν ε, αυτές οι γονικές άδειες από μέτρα που θα προστατεύουν από κάθε κατάχρηση τους εργοδότες. Αλλά οι εργαζόμενοι που θέλουν να φροντίσουν ένα μέλος της οικογένειάς τους θα πρέπει και αυτοί να προστατευτούν για να μην αποχωρήσουν από την εργασία. Διευκρινίζω ότι η κατάσταση των ε, μονογονικών οικογενειών δεν λαμβάνεται σχεδόν καθόλου υπόψη από την ε, Κομισιόν. Εγώ θεωρώ ότι η διάρκεια της γονικής άδεια ε, για τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να μπορεί να διπλασιαστεί. Και το ίδιο πρέπει να ισχύει για ε, τους ε, γονείς που πρέπει να φροντίσουν ένα παιδί που έχει μία αναπηρία ή αν υπάρξει υιοθεσία. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Θέλει κανείς το λόγο. Η κυρία Εσταράς. Ευχαριστώ. Σύμφωνα με την πρόταση της κυρίας Μπερζερόν, πράγματι, πρόκειται για μια οδηγία προσαρμογής ε, του πλαισίου αδειών ε, και διευκόλυνση της, ε, του συνδυασμού οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής προσαρμόζοντας το πλαίσιο αυτό στην σημερινή πραγματικότητα. Οι διατάξει αυτές θα επιτρέψουν στους ε, άντρε να αναλάβουν ένα μεγαλύτερο τμήμα των οικογενειακών ευθυνών. Ε, μειώνοντας τις, ε, διαφορές, διαφορές, ε, λαμβάνοντας ε, μέτρα για την προσαρμογή των μητρικών και πατρικών αδειών, διευκόλυνση των ατόμων που φροντίζουν κάποια ασθενή, κάποιους ασθενείς ηλικιωμένους κλπ. Στην αιτιολογική σκέψη 4 για τη σήμαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία υπάρχουν κάποια ζητήματα. Ε, είναι πολύ καλό το νέο αυτό. Ε, και μετά η προστασία εναντί απολύσεων και το βάρος απόδειξη γι' αυτό ε, σε περίπτωση απόλυσης ε, ατόμου που έχει ζητήσει άδεια, αναρωτική άδεια. Ε, επίσης ε, είναι πολύ καλό που γίνεται δήλωση σεβασμού της αρχής της επικουρικότητας. Ε, Επί της ουσίας ε, μιλούμε για θέματα απασχόληση. Εγώ είμαι μέλος της Επιτροπής Γυναικών και προσπαθούμε να προσαρμόσουμε το νομοθετικό πλαίσιο στην πραγματικότητα ε, με εγγύηση της εφαρμίσης της ε, αρχής της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών προκειμένου και τα δύο φύλλα να έχουν τις ίσες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τη θετική μου γνώμη σε σχέση με την εργασία της κυρίας Μπερζερών και τη συμβολή που θελήσαμε να κάνουμε στην υποβολή κάποιων, με την υποβολή κάποιων τροπολογιών ε, αφορά κάποια σημεία που και η ίδια ανέφερε ώστε να μπορέσουμε να οθήσουμε λίγο πιο πέρα το σώρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όπως έλεγε συνάδελφος να στηρίξουμε την ε, αντιπαράθεσή μας σε οποιαδήποτε διάκριση που να βασίζεται στο φύλλο, να προωθήσουμε τη συνδυασμό επαγγελματικής με οικογενειακή ζωή και να εμποδίσουμε την αναχέ, την, ε, τον αποκλεισμό των γυναικών από την κοινωνική ε, και επαγγελματική ζωή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λεμπρετών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το κείμενο είναι προφανώς ενδιαφέρον γιατί μας επιτρέπει να σημειώσουμε πρόοδο στο, σε θέματα ισότητας ανδρών και γυναικών επιτρέποντας τους αντρές ε, να παίρνουν πιο εύκολα άδειες είτε μικρής ε, άδεια ε, πατρικές ε, άδειες πατρότητα, συγγνώμη, ε, είτε γονικές άδειες, ε, προφανώς είναι πολύ καλό. Απ' την άλλη μεριά να σας πω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσονται αυτά τα κοινωνικά δικαιώματα. Αυτό δεν έχει άμεση σχέση με το ίδιο το κείμενο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προσπαθεί να δείξει ότι φροντίζει τα κοινωνικά δικαιώματα. Από την άλλη μεριά ακολουθεί μια υπερφιλελεύθερη οικονομική πολιτική ε, που πλήττει τα κοινωνικά δικαιώματα. Θα πρέπει ε, και να κάνουμε το καθήκον μας βέβαια και να υπενθυμίζουμε την πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Thank you very much. Any other Πρόεδρος, θα ήθελε κανείς άλλο το λόγο. Όχι. Κομισιόν. Ευχαριστούμε πολύ την ε, κυρία Μπερζερόν και όλα τα μέλη για τα καλά τους σχόλια. Είμαι η Εφη Αναστασίου από την Γενική Διεύθυνση ΕΜΠΛ. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες των διαφόρων τροπολογιών. Η ίδια η κυρία Μπερζερόν ε, εστίασε κυρίως στην γονική άδεια Οπότε αυτό θα σχολιάσω και εγώ καταρχήν. Να πω βέβαια ότι βασικός στόχος αυτής της πρωτοβουλίας ε, είναι να αντιμετωπίσουμε το θέμα της υποεκπροσώπησης των γυναικών στην αγορά εργασίας. κυρία Μπερζερόν πολύ σωστά παρουσίασε τις προκλήσεις. Να υπογραμμίσω όμως εγώ πόσο σημαντικό είναι να δώσουμε βάρος και στο ρόλο των ανδρών Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας προσπαθούμε να διευκολύνουμε και να ενθαρρύνουμε τους άντρες να αναλάβουν ένα πιο δραστήριο ρόλο στα οικογενειακά βάρη. Η γονική άδεια βέβαια είναι το βασικό κομμάτι αυτής της οδηγίας, αυτής της πρωτοβουλίας. Ήδη φύσταται ως δικαίωμα αλλά στην ε, ισχύουσα οδηγία γονικής άδειας ε, ε, δεν υφίσταται ιδιαίτερη ενθάρρυνση προκειμένου κάποιο να παίρνει, να και να παίρνει αυτή την άδεια οπότε θέλουμε να ενισχύσουμε αυτό το δικαίωμα προκειμένου άντρες και γυναίκες να μοιράζονται πιο ισότιμα τους ρόλους. Θα πρέπει να πάρουμε υπόψη όλους, όλες παραμέτρους από κοινού μαζί γιατί ε, υπάρχουν κράτη-μέλη που έχουν γονικές άδειες που δεν πληρώνονται ε, ε, τις οποίες συνήθως δεν παίρνουν οι άντρες ή αν δεν επιτρέπεται ακόμα όμως και αυτές που πληρώνονται και επιτρέπονται ε, συνήθως οι άντρες τις μεταφέρουν στις γυναίκες τους. Θέλουμε ε, απ' την άλλη μεριά, να εξασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες δεν, δεν θα μένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα εκτός αόρας εργασίας. Συνεπώς, η αύξηση του, των, των ημερών άδεια ε, και η μη δυνατότητα μεταφοράς θα σημαίνει ενδεχομένως ότι οι γυναίκες θα μένουν περισσότερο χρόνο εκτός αγοράς εργασίας. Επίση, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις, ε, με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπίσουμε και τις μεγάλες μισθολογικές και συνταξιδοτικές διαφορές. Ε, μετά, οι ε, αναρωτικές άδειε που πληρώνονται είναι σημαντικό να αφορούν και τους ε, και να είναι σε υψηλό επίπεδο η αμοιβή. η πρόταση είναι στο 50% του μισθού, όμως ε, επιθεωρούμε ότι δεν είναι πολύ ψηλό, αρκετά υψηλό. Ε, αν ε, η αναρωτική άδεια πληρώνεται στο 50% του μισθού, δεν θα είναι αρκετό για να ζητά κάποιος την αναρωτική άδεια όταν τη χρειάζεται. Ένα άλλο θέμα, το οποίο αφορά τους μόνους γονείς. Ο στόχος είναι οι γυναίκες, όπως είπα, να μην μένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα εκτός αγοράς εργασίας. Οπότε λαμβάνουμε υπόψη ότι οι μόνοι γονείς είναι συνήθως στις περισσότερες περιπτώσεις γυναίκες. Αν διπλασιάσουμε την γονική άδεια, αυτό θα σπρώξει τις γυναίκες ακόμα μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα εκτός ε, αγορά Βέβαια αναγνωρίζουμε ότι οι μόνε γυναίκε χρειάζονται στήριξη Γι' αυτό και έτσι κι αλλιώ η οδηγία καθορίζει τα ελάχιστα δικαιώματα, τα κράτη-μέλη μπορούν να τα διευρύνουν αν το επιθυμούν. Προτείνει η Κομισιόν λοιπόν, αντί να επιμικίνουμε τις γονικές άδειες για τους μόνους γονείς, να τους δώσουμε πρόσθετα δικαιώματα τα οποία θα τους στηρίξουν ε, και αποφύγουμε έτσι την ε, διατήρηση των γυναικών εκτός της αγοράς εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you as well. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Η συγκήτρια θα ήθελε να πει κάτι αυτή τη στιγμή. Δύο λόγια μόνο. Στον κύριο Κασπαρακ να πω ότι ακριβώς ε, βρισκόμαστε στην ε, ίδια κατεύθυνση. Ε, επί της αρχής. Η γονική άδεια για τους άντρες ε, είναι πιο πολύ φιλοσοφικό θέμα, δεν αφορά μόνο τα χρήματα. Θα πρέπει να καταλάβουν οι άντρες ότι είναι και αυτοί απαραίτητοι για την αντροφή του παιδιού τους. Δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουν την γονική ε, άδεια ως ένα τρόπο να μεταφέρουν περισσότερα δικαιώματα στις γυναίκες τους πράγματι μια γονική άδεια θα μπορούσε να υποσκάψει την οικονομική σταθερότητα του, της οικογένειας. Θα πρέπει να το προσέξουμε. Ε, τώρα, οι γυναίκες που εργάζονται και φροντίζουν έναν ηλικιωμένο ε, ένα ηλικιωμένο άτομο. Εγώ το έκανα, ε, ο άντρας μετανάστης, για 25 χρόνια. Και εγώ εργαζόμουν και τον φρόντιζα. Ε, εγώ ήμουν επικεφαλής επιχείρησής μου και μπορούσα να, να το κάνω αυτό εύκολα. Ε, αλλά αν, δεν, αν ήμουν απλός υπάλληλος θα ήταν πολύ δύσκολο να κοιμηθώ στις 2 το πρωί και την επόμενη μέρα να ξυπνήσω να πάω στη δουλειά μου. Ε, μιλώ βέβαια εδώ για τους συζύγους αλλά έχουμε και παιδιά που είναι ανάπηρα κλπ. Ε, και έχω την εντύπωση ότι αυτό το πρόβλημα το, το είδαμε λίγο πρόχειρα. Κατά τα άλλα, ε, συμφωνώ με όλες τις τροπολογίες που υποβάλλατε σε ό,τι αφορά την ε, γονική άδεια. οι τροπολογίες μπορούν να υποβληθούν μέχρι 23 Νοεμβρίου. Αυτή είναι η προθεσμία. Ευχαριστώ και τα ξαναλέμε. Thank you very much. Πρόεδρος. Η προθεσμία υποβολή τροπολογιών, επαναλαμβάνω και εγώ, είναι 23 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. ...24 Νοεμβρίου. 24 Νοεμβρίου το μεσημέρι. Περνάμε στο σημείο 25. Έκθεση απαλλαγής 2016, Γενικός Προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δικαστήριο. Εισηγητής είμαι εγώ ο ίδιος, οπότε να υπογραμμίσω τα εξή σημεία της έκθεσης. Σημείο 2. Ο προπολογισμό του δικαστηρίου είναι καθαρά διοικητική φύσεως. Ε, το 75% περίπου του προπολογισμού δαπανάται για τα πρόσωπα που συνδέονται και εργάζονται στο δικαστήριο και τα υπόλοιπα ε, και, για, τα, και για άλλες δαπάνες. Η έκθεση υπογραμμίζει ότι το 2016 το ελεγκτικό συνέδριο δεν εξέδωσε ειδική έκθεση για το δικαστήριο. Θα θυμάστε ότι το ζητήσαμε το ελεκτικό συνέδριο να υποβάλει ε, έκθεση για το δικαστήριο αλλά για το 2017 ενώ η έκθεσή μου αφορά το έτος 2016 αυτό ήθελα να το διευκρινίσω. Και το σημείο 7 της έκθεσης ε, εκφράζει την ικανοποίησή μας για το γεγονό ότι το δικαστήριο καταβάλει προσπάθειες για την ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων. Αυτά είναι βασικά αυτά που ήθελα να πω εγώ. Η κυρία Ντελβό θα ήθελε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ε, πρόταση έκθεσης. Δεδομένου ότι αύριο θα συναντηθούμε με τους ε, δικαστές του, του δικαστηρίου, θα μπορέσουμε και εκεί να ανταλλάξουμε απόψεις. Στο σημείο 7 θα ήθελα να σχολιάσω το εξής. Πιστεύω ότι είστε υπερβολικά ε, θετικό σε σχέση με τις προσπάθειες που έχουν γίνει για την ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων. Με 7 συνολικά γυναίκες στο δικαστήριο ε, είμαστε ακόμα πολύ μακριά από την ισότητα. Και άλλωστε δεν είναι το δικαστήριο που κάνει τις προσπάθειες, τα κράτη-μέλη προτείνουν τους υποψηφίους. Το δικαστήριο δεν έχει να πάρει κάποια απόφαση εκεί, οπότε θα υποβάλω μια τροπολογία σε αυτό. Κομισιόν. Όχι. Ε, η προθεσμία υποβολή τροπολογιών η 4η Δεκεμβρίου το μεσημέρι. Σημείο 26. Έκθεση αποστολής μετά την επίσκεψη της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων στην Silicon Valley. Όπως γνωρίζετε, ε, για λόγους που με ξεπερνούσαν δεν κατάφερα να συμμετάσχω στην αυτή, σε αυτήν την αποστολή, οπότε θα δώσω το λόγο στην κυρία Γκέριγκερ που ήταν επικεφαλής της ε, αντιπροσωπής ως πρώτη αντιπρόεδρος. Ε, σας ευχαριστώ. Ήθελα να σας κάνω μια σύντομη έκθεση ε, για την επίσκεψη που έλαβε χώρα ανάμεσα στις 30 Οκτωβρίου και στις 2 Νοεμβρίου. Τα μέλη αυτής της Επιτροπής Μετέβησαν στο Σαν Φρανσίσκο και μπορέσαμε να έρθουμε σε επαφή με διάφορους εταίρους αλλά και επιχειρήσεις εκεί. Επιχειρήσεις που εργάζονται στην Silicon Valley. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη. Να σας θυμίσω ποιοι συμμετείχαν εξ ονόματος της Επιτροπής μας από το ΕΛΚ ο κύριος Φως και ο κύριος Σβιέπκα για τους σοσιαλιστές η κυρία Κάουφμαν και εγώ εξ ονόματος του ΙΣΙΑΡ ο κύριος Καρίμα η κυρία Ρέντα από τους Πράσινους, η κυρία Μπερζερό ε, από το FTD ε, και είχαμε επίσης μαζί και τον κύριο Έλερ που είναι ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας για τις ε, σχέσεις και τη συνεργασία με τις ΕΠΑ. Είχαμε 13 ε, συναντήσεις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, ήταν πολύ εντατικό δηλαδή το πρόγραμμά μας, εντατικό μεν αλλά ενδιαφέρον. Ε, νομίζω πως αποκομίσαμε πολλά, καθώς κοιτώ για δυόμιση μέρες ε, ε, συνεδριάσεων, συνεδριάσεων εξαιρετικά ενδιαφερόντων. Τα μέλη αυτής της Επιτροπής, όπου πήγαν μαζί με μένα, φαντάζομαι ότι θα προσθέσουν κάποια λόγια. Στις 30 Οκτωβρίου Μόλις στάσαμε, συναντήσαμε εκπροσώπους επιχείρησης Sky Venture. Τις επόμενες μέρες συναντήσαμε εκπροσώπους της 21st ε, Century Fox, της Universal Music, της Skyled, επίσης εκπροσώπους του Facebook, του Electronic Foundation, της Google, της Apple. Ε, επισκεφθήκαμε το Πανεπιστήμιο του Stanford Είδαμε εκπροσώπους της Walt Disney, της Pixar, της Cisco System. Ε, επισκεφθήκαμε τον Οργανισμό ευρεστεχνιών του ΙΠΑ ε, στο Σαν Χωσέ και επίσης ε, νόσεις των νεοφιών εταιριών καθώς και εκπροσώπους μιας νέας εταιρείας που μας διηγήθηκε την εμπειρία του. και κυρίως επικεντρώθηκε στα θέματα που μας ενδιαφέρουν, δηλαδή στην οικοδόμηση της ενιαίας, αγοράς, της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Μιλήσαμε, ας πούμε, για δικαιώματα πνευματικά, ε, ε, για σήματα κτλ. Όλα αυτά που μας ενδιαφέρουν ε, συζητήθηκαν. Ε, μπορείτε να με προσέξετε λίγο, παρακαλώ. Οι τρεις εκεί πίσω, μήπως μπορείτε να συζητήσετε αλλού, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Είχαμε την ευκαιρία να συγκρίνουμε τις απόψεις μας για το θέμα των παραβιάσεων των ε, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο ίντερνετ. Ε, ε, είδαμε πώς θα λειτουργήσουν στο μέλλον ορισμένες ανακαλύψεις καινοτομίε που σχετίζονται με την τεχνητή ευφυΐα ή τα αυτόνομα αυτοκίνητα και πάντοτε όλα αυτά υπό το φως του δικαίου, του, ε, του δικαίου που καλύπτει τα πνευματική ιδιοκτησία και το σεβασμό του δικαίου. Τέλος, να σας δώσω το παράδειγμα μιας άποψης που θεώρησα ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, συναρπαστικό και ε, προέρχεται από το Ίδρυμα Electronic Frontier. Μα έδειξαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, μάλιστα και η μέρα του Halloween ορισμένοι από του υπαλλήλου, ήταν ήδη μεταφιεσμένοι για να γιορτάσουν ε, το Halloween μετά από την συνάντηση μαζί μα. αλλά αυτό που θέλω να σα πω είναι το εξή. Ρωτήσαμε πώ μπορούσαμε να καταφέρουμε να μην γίνονται παραβιάσεις των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο ίντερνετ. Και ήταν πολύ απλή. Είπαν αρκεί να μετατρέψει το ίντερνετ σε κάποιο είδος καλωδιακής τηλεόρασης, όπου δεν υπάρχει πρόβλημα με τα πνευματικά δικαιώματα. Αν όμως θέλουμε το ίντερνετ να μείνει ένα ελεύθερο, ένας ελεύθερος ανοιχτός χώρος, ε, όπου θα γίνονται οι συναλλαγές και θα προωθούνται οι συναλλαγές και όπου δεν μπορούμε να μεταχειριστούμε και να αντιμετωπίσουμε όλους τους δημιουργούς με τον ίδιο τρόπο, τότε το ίντερνετ θα μπορέσει να δημιουργεί να, λειτουργήσει ως μια τεράστια ε, μηχανή, μηχάνημα φωτοτυπικό όπου ε, θα μπορεί να μεταφέρεται το υλικό χωρίς να αμείβονται οι δημιουργοί και οι δημιουργοί δεν, δεν εξοργίζονται πάντοτε ε, τη στιγμή που κάπως πληρώνονται. μιλάμε για την χρηματοποίηση, την απόδοση των χρημάτων σε κάθε στιγμή. Αυτά έχω να σας πω. Ο συνάδελφος Φως. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για αυτή την παρουσίαση της επίσκεψής μας. Καταρχάς θέλω να επενέσω ιδιαίτερα τη γραμματεία. Η γραμματεία τα οργάνωσε και τα προτίμασε όλα θαυμάσια και επίσης ε, ε, κατά την επίσκεψη μας βοήθησε όμως ε, να κάνω μια σύσταση. Ε, αν ξαναπάμε, ίσως θα μπορούσαμε να μείνουμε λίγο περισσότερο στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Αυτή μόνο μία ώρα που κάναμε, που τους είδαμε, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Θα μπορούσαμε να έχουμε μείνει λίγο περισσότερο. Ε, κατά τα άλλα ήταν πολύ πυκνό πρόγραμμα. Περίχε πολλά θέματα, ήδη αναφέρθηκαν και επίσης ε, είδαμε και μία μη κυβερνητική οργάνωση αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι ε, δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί η κατάσταση έτσι όπως είναι. Δεν είναι μόνο παραβίαση ε, των ιδιωτικών δεδομένων, είναι και προσβολή ατόμων που γίνεται στο ίντερνετ. Εμείς ε, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό ε, να ε, τηρούνται οι αξίες μας. Δεν είναι να το να λέμε «Ε, καλά ίντερνετ είναι, ας γίνει ό,τι να είναι». Θα ήταν λάθος αυτό να το δεχθούμε λοιπόν. Αλλά κατά τα άλλα ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι συζητήσεις που κάναμε. Πολύ ενδιαφέρον να δούμε επίσης πώς οι επιχειρήσεις αυτές σχετίζονται με τις πλατφόρμες και πώς από την άλλη μεριά πώς αυτές οι πλατφόρμες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα νομικά θέματα που τίθενται κάπως καλύτερα. Πρέπει όλα αυτά να συνδυαστούν καλύτερα. Ήταν λοιπόν θαυμάσιο αυτό ότι σε όλες τις συζητήσεις που κάναμε ε, είχαμε συζητήσεις υψηλού επίπεδου και σας ευχαριστώ και άλλη, επίσης ε, άλλη μια φορά. Ναι, ναι. Ε, ιδίως συμφωνώ με αυτό που είπατε ότι πρέπει να ξαναπάμε. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κάουφμαν. Βεβαίως, ευχαρίστω. Φτάνει ο πρόεδρος μας να έχει διαβατήριο που να ισχύει. Τότε θα μπορούσαμε να ξαναπάμε. Ευχαριστώ πολύ και εγώ τη γραμματεία. Όντως ήταν πολύ πυκνό το πρόγραμμα και κουραστικό θα έλεγα. Και από πλευράς περιεχομένου βρήκα πολύ ενδιαφέρουσες για πολύ διαφορετικούς λόγους τις συναντήσεις. Μάθαμε πώς αντιμετωπίζουν τα θέματα εκεί, είδαμε τις απόψεις τους. Για το ίντερνετ. Το θέμα είναι το ίντερνετ όπως και ο πραγματικός κόσμος πρέπει να τηρούν το δίκαιο. Το θέμα όμως είναι πώς εφαρμόζεται. Πρέπει να το δούμε περαιτέρω. Αναφέρθηκαν μια σειρά θέματα όπου είπα «Α, ενδιαφέρον, πρέπει να το σκεφτώ». Δηλαδή, εγώ από αυτές τις ε, συζητήσεις ε, μου δημιουργήθηκαν περισσότερες ερωτήσεις. Βεβαίως, ε, Καταλαβαίνω ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε αναλυτικά πρακτικά για κάθε συνάντηση, αλλά θα ήθελα να παρακαλέσω τη Γραμματεία αν θα μπορούσε να συνοψίσει κάπως το περιεχόμενο των συναντήσεών μας. Ξέρω ότι έχει πολύ δουλειά η Γραμματεία, αλλά νομίζω ότι θα μας βοηθούσε να έχουμε μια συνόψηση. Να ξαναδούμε δηλαδή τι υπόθηκε στις συναντήσεις αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος. Ναι, θα υπάρξει μια έκθεση για την ε, αποστολή αυτή. Ο κύριος Βίφκα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ συμφωνώ με τις ευχαριστίες ε, προς τους συναδέλφους της Γραμματείας που ε, ε, προετοίμασαν θαυμάσια αυτή τη συνάντηση και συμμερίζομαι και τις απόψεις των συναδέλφων. Αλλά να προσθέσω και εγώ μερικές δικές μου σκέψεις. η διαφορά προσέγγιση όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών εξακολουθεί να είναι ένα χάσμα. Υπάρχει απόλυτη απόκληση. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν μπορούμε κάπως να επιχειρήσουμε να συγκλίνουν οι απόψεις μας. Για παράδειγμα, όταν είδαμε το Facebook, συζητήσαμε το θέμα της ευθύνης για το περιεχόμενο που αναρτάται για παράδειγμα αυτοί που διαχειρίζονται από πλευράς Facebook ε, τις αναρτήσεις πώς μπορεί να αποφασίσουν ότι κάποια περιεχόμενα είναι παράνομα ή ότι ξεπερνούν κάποια όρια και κάποιους κανόνες υπάρχουν διαδικασίες λοιπόν αλλά είναι υποσυνεχή ε, τροποποίηση για να ε, συμμορφούνται προς το δίκαιο και τις αξίες μας γιατί καμιά φορά είναι και παράνομα αυτά που γράφονται και ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπαν και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Οι επιχειρήσεις βεβαίως αντιμετωπίζουν νομικά θέματα. Και ξέρετε ότι οι νομομαθείς μπορεί επίσης να εκπροσωπούν διαφορετικά συμφέροντα. Τους παραγωγούς, τους παρόχους υπηρεσιών, τους δημοσιογράφους, τους ε, ε χρήστες και για πολύ διαφορετικά θέματα και τομεί. Μπορούμε λοιπόν να διαφωνούμε, ορισμένα πράγματα μπορεί να μα αρέσουν, αυτό είναι το ένα, αλλά πρέπει να μην ξεχνάμε ότι ε, πρέπει να δούμε και ποια είναι τα συμφέροντα της δικής μας αγοράς. Πώς θα σεβαστούμε εμείς τη δική μας αγορά, πώς θα εφαρμόσουμε τις αξίες μας, πώς θα ενθαρρύνουμε τους Αμερικανούς να δεχτούν τις δικές μας απόψεις. Εν πάση περιπτώσει, αυτέ οι επισκέψει πιστεύω ότι πρέπει να γίνονται τακτικά, γιατί πραγματικά διευρύνει τους ορίζοντές μας μια τέτοια επίσκεψη, Μα επιτρέπει να λάβουμε υπόψη άλλες απόψεις. Θεωρώ ότι η ζουρή επιτέλους κατάφερε, επιτέλους, να πείσει τα αρμόδια όργανα του Κοινοβουλίου ότι πρέπει να γίνονται τέτοιες επισκέψεις και θεωρώ ότι και στο μέλλον θα έπρεπε ακριβώς να απαιτήσουμε εκ νέου τέτοιες επισκέψεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θέλω να κάνω ακόμα μια παρατήρηση. Όχι ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας, αλλά ως μέλος της αντιπροσωπείας θα ήθελα να πω ότι είδαμε αυτόματα αυτοκίνητα, αυτόνομα με συγχωρείτε, χωρίς οδηγό δηλαδή. Και αναρωτηθήκαμε ποιος θα φέρει την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος. Ο οδηγός είναι ανύπαρκτος σε αυτά τα αυτοκίνητα. Και η απάντηση ήταν ότι σε περίπτωση ατυχήματος οι Αμερικανοί δεν σκέφτονται να δημιουργήσουν ένα νέο δικαίωμα που θα συνδέεται με τα ρομπότ ή με την τεχνητή ευφύεια. Και μας είπαν πάνω κάτω, ας περιμένουμε το πρώτο και βλέπουμε. Τότε θα προχωρήσουμε και θα έχουμε τις πρώτες υποθέσεις. Ε, η κυρία Δηλυβόμος όμως είπε ότι θα έπρεπε η ευθύνη να, να τη φέρει αυτός ο οποίος έχει φτιάξει το αυτοκίνητο ή έχει ε, φτιάξει το λογισμικό, αλλά υπάρχει και η πτυχή του ίντερνετ, γιατί έχουμε δορυφόρους ε, μέσω των οποίων γίνεται η οδήγηση. Η απάντηση λοιπόν δεν είναι τόσο εύκολη. Δεν είναι τόσο απλή. Και Τέλος. Ακούσαμε ότι όταν λείπει το ίντερνετ συχνά μένουμε απ' έξω. Όταν δεν έχουμε ένα κινητό μένουμε απ' έξω. Οπότε είναι δύσκολα. Αυτό μου θυμίζει την αποστολή μας στο Λουξεμβούργο στην υπηρεσία μετάφρασης, εάν θυμάστε, όπου η υπηρεσία μετάφρασης μας έδωσε μια εικόνα της εργασίας της, αλλά δεν έχει μεταφραστεί λόγω του κόστους. Ε, so, ε, ε, συνεχίζουμε με το σημείο 27. Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις ενέργειες οι οποίες προέβη η Επιτροπή μετά το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ε, ρομποτική. Ο λόγος στην κυρία Ντελβό. Μας απομένουν μόνο 12 λεπτά δυστυχώς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Το θέμα αυτό είναι στην ημερήσια διάταξη για να δούμε τι έχει συμβεί από το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μετά το οποίο έλαβε χώρα στην Ολομέλεια το Φεβρουάριο. Λάβαμε την απάντηση της Κομισιόν, της, Ε, η Επιτροπή πολύ ευγενικά μας είπε ότι ήταν πολύ καλή εκθεσή μας και ότι σε γενικές γραμμές συμμερίζεται τις ανησυχίες μας. Ε, δεν έχει όμως να κάνει κάτι, ε, να ανακοινώσει κάτι πολύ συγκεκριμένο γιατί αυτή τη στιγμή εξετάζει το ζήτημα. Γίνονται εσωτερικέ διαβουλεύσει και βέβαια είναι και πολύ περίπλοκο το θέμα. Η τεχνολογία από την άλλη μεριά προοδεύει πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε ε, δεν είναι δυνατόν ακόμα να ληφθούν αποφάσεις, να υποβληθούν προτάσεις για νομοθετικά κείμενα ε, τα οποία ενδεχομένω θα μπορούσαν να περιορίσουν ή να καθυστερήσουν την εξέλιξη, την τεχνολογική εξέλιξη ή την καινοτομία. Θα ήθελα από την άλλη μεριά εγώ να πω τα εξή. Ε, εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό η Κομισιόν να υποβάλει πρόταση ό,τι αφορά την νομική ευθύνη σε περίπτωση βλάβης τρίτων. Για παράδειγμα, ε, αυτοκίνητα χωρίς οδηγό. Δεν βρισκόμαστε βέβαια στο επίπεδο 5, αλλά ε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε επιστάδιο δοκιμών ε, και υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία ήδη νομοθετούν για το ζήτημα. Οπότε το δικό μας επιχείρημα ήταν ότι να μια φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να καθορίσει αρχές που θα εφαρμοστούν αργότερα από όλα τα κράτη-μέλη. Αν Ε, δεν διαθέτουμε τέτοιου είδους αρχές εξ αρχής, θα χρειαστεί να περάσουμε τά ε, διορθωτική νομοθεσία αργότερα. Η Κομισιόν είναι εδώ παρούσα, οπότε μπορεί να μας δώσει ενδεχομένως κάποιες ε, απαντήσεις σε αυτά. Γιατί, γιατί η Κομισιόν έχει ήδη κάνει διαβουλεύσεις, ε, και μελέτες δεν μπορώ να πω ότι έχω κάποιες προκαθορισμένες ιδέες, αλλά θα ήθελα να ακούσω την Κομισιόν για αυτό το ζήτημα. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ηθικής και των προτύπων και προδιαγραφών των μπορούμε να πρωτοπορήσουμε στην Ευρώπη και να καθορίσουμε συγκεκριμένες ε, αρχές για την αυτοκινητοβιομηχανία. Ε, διάβασα με ενδιαφέρον την πρόταση του πρόεδρου Μακρόν περί μιας ε, υπηρεσίας καινοτομίας και η ε, τεχνητή νοημοσύνη σίγουρα θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο αυτής της υπηρεσίας. Και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, έχουμε, μια ακρόαση για τη, τα ρομπότ, τη ρομποτική. Η τελική έκθεση δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα. Ενώ η Υπερές ε, έχει κάνει μια μελέτη για τα αυτόνομα αυτοκίνητα, ούτε από εκεί όμως έχω νέα. Όπως και, για την ακρόση, και από την ακρόση για τα ε, αυτόνομα αυτοκίνητα. Ίσως λοιπόν θα μπορούσαμε να προσπαθήσουμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα από αυτές τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναλυθεί. Τέλος, διαπιστώνω με ε, σχετική ικανοποίηση ότι το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, στα συμπερασματά του συμπεριέλαβε ε, μία παράγραφο για την τεχνητή νοημοσύνη δια της οποίας ανακοινώνεται ότι τα κράτη-μέλη αναμένουν μία σύσταση κάποιο, κάποιο κείμενο της Κομισιόν, κάποια πρόταση της ενδεχομένως για το θέμα αυτό. Εδώ σταματώ για να μην μονοπολίσω τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Κύριο Άντερσον. Θα μιλήσω μετά την Κομισιόν. Ωραία. Η Κομισιόν. Καλή σας μέρα. Ονομάζομαι Χέκυλα από την Γενική Διαμτσή Κόνεξ, επικεφαλής της, ε, της μονάδας ρομποτικής και τεχνητής νομοθεσίνης. Για τα πιο νομικά θέματα θα αφήσω άλλου συναδέλφου να μιλήσουν, αλλά να σα πω τα εξή. Ήδη εργαζόμαστε σε αυτό το, επί αυτού εδώ και αρκετό καιρό. Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα και πιστεύουμε ότι το ψήφισμά σας ήταν πολύ χρήσιμο γιατί μας στήριξε σε πολλά θέματα, μας έδωσε επιχειρήματα για να κινηθούμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Έτσι ώστε να δούμε το ζήτημα από την ευρωπαϊκή οπτική γωνία. Συμφωνώ βέβαια με το ότι υπάρχει ανάγκη να ακολουθεί μια ευρωπαϊκή προσέγγιση. Γιατί, γιατί τα διάφορα μεμονωμένα κράτη-μέλη δεν μπορούν από μόνα τους να κάνουν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι μόνο θέμα νομικής υφής. Και δεν πρόκειται καν μόνο για θέμα κατακαιρματισμού από των νομικών πτυχών. Είναι κατά κύριο λόγο θέμα έρευνας και βιομηχανικής ισχύω που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε έχουμε και τις δύο αυτές πτυχές που πρέπει να δούμε. Βέβαια, τα κράτη-μέλη μπορούν να νομοθετήσουν και σε μερικές περιπτώσεις το κάνουν, όπως στο θέμα των αυτόνομων αυτοκινήτων ελέγχθη αυτό, ούτε μπορούμε να το αποφύγουμε. Όμως εργαζόμαστε πολύ εντατικά εξετάζοντας την, ε, ε, τα, τις ηθικές πτυχές, τις οικονομικές πτυχές, τις βιομηχανικές πτυχές, τις νομικές πτυχές, τις κοινωνικές πτυχές, τις τεχνολογικές πτυχές. Ε, είμαστε σε επαφή με την κοινωνία των πολιτών και μην ξεχνάτε ότι την επόμενη εβδομάδα ξεκινά η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ρομποτικής πολλές ε, εταιρείε ε, και εργαστήρια θα ανοίξουν, θα δείξουν, θα επιδείξουν τις, ε, τα σχέδιά τους και τα πρωτότυπά τους. Στο επόμενο πρόγραμμα του Horizon 2020 έχουμε σχέδια έτσι ώστε όλα αυτά τα προγράμματα και τα προϊόντα να γίνουν πιο προσβάσιμα, να εκδημοκρατιστεί σε εισαγωγικά ο τομέας αυτός, έτσι ώστε να ε, παρουσιαστεί ενώπιον της κοινωνίας. Πρέπει να πρωτοπορήσουμε για να βασιστούμε στις αρχές μας, διότι αλλιώς τα ίδια πράγματα θα τα κάνουν κάποιοι άλλοι βασιζόμενοι στις δικές τους αρχές. Ε, προετοιμάζουμε διάφορα πράγματα, διάφορες πρωτοβουλίες. Θα απαντήσουμε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου καταρχήν. Ακόμα και αν δεν μας το είχε ζητήσει το Συμβούλιο θα το επράταμε, θα υποβάλουμε κάποιο κείμενο για μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στην ε, τεχνητή νοημοσύνη. Θα ανταποκριθούμε λοιπόν εν ευθέτω χρόνο για το θέμα, για τα ηθικά ζητήματα προκύπτουν, τα ζητήματα δεοντολογίας, ε, προφανώς γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή υφίστανται πολλές διεθνείς πρωτοβουλίες. Οπότε τίθεται ερώτημα αν θα πρέπει να ακολουθήσουμε και εδώ μια ευρωπαϊκή προσέγγιση, αν θα ακολουθήσουμε μια παγκόσμια προσέγγιση. Δεν είναι εύκολο να απαντήσουμε σε αυτό το ζήτημα. Είναι και αυτό ένα κομμάτι της εργασίας μας. Οπότε Αυτά από την πλευρά μου να αφήσω και κάποιους συναδέλφους να μιλήσουν. Δυστυχώς έχουμε πολύ περιορισμένο χρονικό οριζόντα. Μία μόνο φράση για την οδηγία ελαττωματικών προϊόντων. Ε, πράγματι ε, συνεχίζεται η αξιολόγηση με τους ε, εμπλεκόμενους φορείς και ενδιαφερόμενους και λαμβάνουμε υπόψη και την κλαδική νομοθεσία όπου υπάρχει. Για παράδειγμα την οδηγία περί μηχανισμάτων. Όλα αυτά θα τα συνδυάσουμε με συμπεράσματα από τα οποία έχετε ήδη εσείς, τα οποία έχετε εσείς δημοσιεύσει, προκειμένου να εντοπιστεί πώς θα απονέμονται οι ευθύνες ε, Ε, κατόπιν και τη ε, απέτηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να ακολουθήσουμε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση. Ο τρίτος Είμαι ο τρίτος εκπρόσωπος της Κομισιόν από την Γενική Διεύθυνση Justice. Ε, μας ενδιαφέρουν τα ιδεοντολογικά ζητήματα και τα ζητήματα ε, αποζημιώσεων και ευθυνών. Συνεργαζόμαστε με τους ε, συναδέλφους της Connect και της Grow. Ε, να σας πω ότι ήδη εργαζόμαστε για θέματα ευθύνης ε, και είχαμε ήδη μια ανακοίνωση πριν το ψήφισμα του Κοινοβουλίου δύο ε, ε, ε, διαβουλεύσεις και ένα εργαστήριο μέσα στο καλοκαίρι στο οποίο ήταν παρούσα η κυρία Ντελβό. Οπότε το θέμα της νομικής ευθύνης το εξετάζουμε εμείς στην Κομισιόν από όλες τις πλευρές, από όλες τις γωνίες. Είναι πολύ περίπλοκο θα ανταποκριθούμε, θα απαντήσουμε μάλλον στα αυτά που είπε το Κοινοβούλιο και θα ανταποκριθούμε σε αυτά που μας ζήτησε το Συμβούλιο. Όμως πρέπει πρώτα να εξετάσουμε το ζήτημα σε βάθος. Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να προωθούμε την καινοτομία, να μην την πνίξουμε, ε, διατηρώντας όμως τις αρχές μας, τα θεμελιώδη μας δικαιώματα, την ε, κοινωνικο-οικονομική μας ε, δομή κλπ. Πρέπει λοιπόν να γίνει αυτό, αλλά πρέπει να το κάνουμε καλά, γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε χρόνο. Χαιρόμαστε που μπορούμε να συνεργαστούμε. Περιμένουμε τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης, της έκθεσης για το κόστος της μη Ευρώπης και θα τα λάβουμε υπόψη μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ε, παρακαλώ κύριε Άντερσον με λίγα λόγια. Ναι, Ήθελα να ακούσω την άποψη της Κομισιόν και το έργο της. Ε, εξακολουθώ να είμαι πολύ περίεργος για το τι θα προτείνει η Κομισιόν. Ε, δεν ικανοποιήθηκε η περίεργιά μου. Παρ' όλα αυτά αναμένω με ανυπομονησία τα αποτελέσματα της δουλειάς σας. Ε, να σας... Να πω κι εγώ ότι και εγώ ανησυχώ για θέματα νομικής ευθύνης σε ό,τι αφορά τα αυτόνομα αυτοκίνητα, όπως κύρια Αντελβό. Σε ό,τι αφορά την υπηρεσία, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία είμαι πολύ σκεπτικός ε, για τον πολλαπλασιασμό και την αύξηση του αριθμού των ευρωπαϊκών υπηρεσιών. Όμως, σε αυτή την περίπτωση μπορεί πράγματι να υπάρχουν πολύ καλά επιχειρήματα υπέρ μιας τέτοιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας. Η Κομισιόν Γραπτός μας ε, αναφέρει ότι ε, ε, ε, εξετάζει την δημιουργία μιας, ενός συμβουλίου υψηλού επίπεδου για θέματα ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης. Καλό αυτό. Όμως υπάρχουν θέματα ιδιαίτερα ευαίσθητα πολιτικά και οικονομικά θέματα τα οποία θα πρέπει να επιλύονται επί τη βάση του τι είναι το καλύτερο, το κοινό συμφέρον. Ε, σε, στο παρελθόν, ε, σε τέτοιου είδου συμβούλια ε, έχουμε διαπιστώσει μία μεροληψία υπέρ συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων. Θέλουμε όμως τη συμμετοχή και των επιστημόνων και της κοινωνίας έτσι ώστε οι υπάλληλοι της ε, Κομισιόν να, και θέλουμε μάλλον και οι υπάλληλοι της Κομισιόν να έχουν επαρκείς πόρους ε, και μέσα στη διάθεσή τους για να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Κύριε Φως. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ που τέθηκε αυτό το θέμα στη μέση διάταξη. Καλό είναι αυτό και θα πρέπει να το προωθήσουμε. Και θα έλεγα όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα, γιατί οι τεχνολογικές εξελίξεις ε, καλπάζουν και εμείς ε, βραδιπορούμε με την νομική ε, πλαισίωσή τους. Δεν είναι δυνατόν και πάλι να προχωρήσει η τεχνολογία και εμείς εκ των υστέρων να προσπαθούμε κάτι να διορθώσουμε. Αυτό είναι δύσκολο. Εκ των προτέρων πρέπει να θέσουμε τα ηθικά και νομικά πλαίσια και θα πρέπει να πούμε ότι όποιος αναπτύξει τέτοια προϊόντα θα πρέπει να τηρεί αυτές τις προδιαγραφές. Όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα. Επίσης, Ίσως, ίσως θα έπρεπε να επιδιώξουμε να βρούμε νέους τρόπους, να βγούμε από την πεπατημένη. Γιατί η ψηφιοποίηση ούτως ή άλλως ξεπερνάει όλα τα σύνορα. Γι' αυτό και το νομικό πλαίσιο θα πρέπει να το ξαναδούμε. Να δούμε πώς με άλλες ιδέες, ε, με άλλη διάρθρωση, πώς θα μπορέσουμε να ε, αντιμετωπίσουμε με νέο τρόπο το θέμα και δεν υπάρχει πάντα αυτή η προθυμία κατά τη γνώμη μου για διάφορα θέματα τώρα τελευταία. Αλλά δεν είναι δυνατόν να θεωρούμε ότι οι ίδιες μέθοδοι μπορούν να ισχύσουν για όλα τα θέματα. Αυτό είναι σημαντικό. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που υπάρχουν σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ κύριος Λεμπρετών. Ευχαριστώ πρόεδρε. Τα F.E. ρομπότ εισβάλλουν στη ζωή μας. Είμαστε στο κατόφλι μιας πολύ σημαντικής τεχνολογικής επανάστασης. Άρα πρέπει να το σκεφτούμε το θέμα σοβαρά και να καταλήξουμε σε νομικές λύσεις. Η Επιτροπή βεβαίως που μπορεί να μελέα όσο θέλει χωρίς να μας λέει αυτά που θέλουμε να ακούσουμε, γιατί δεν μας είπαν και πολλά, γιατί όλα αυτά εξακολουθούν να παραμένουν απόρριτα. Στον ένα τον άλλο βαθμό. Ευτυχώς έχουμε το ψήφισμά μας της 16ης Δευτέρου τρέχοντος που προτείνει ορισμένα και να υπογραμμίσω τα εξής δύο. Γιατί αυτό που μου κάνει εντύπωση στις εργασίες μας είναι το πώς μπερδεύουμε το καλό με το λιγότερο καλό. Για παράδειγμα, η καταγραφή των ρομπότ να είναι σε κάποιο μητρό, να μπορούμε να ε, ε, δούμε σε τι αντιστοιχεί το κάθε ρομπότ. Αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Αυτά τα αυτόνομα οχήματα πολύ σύντομα θα περάσουν από μια χώρα στην άλλη. Πρέπει κάπου να είναι καταγεγραμμένα. Μόλις όμως το προτείναμε και είναι λογικό προσθέτουμε θα πρέπει να υπάρξει ένας ευρωπαϊκός ε, ειδικό οργανισμός. Όπως είπε ένας συνάδελφος, αυτός ο πολλαπλασιασμός των ε, ευρωπαϊκών οργανισμών είναι ανισχυτικός. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε ειδικό οργανισμό για τα FE ρομπότ. Και μάλιστα όταν λέω δεν είμαι σίγουρος, εννοώ ότι είμαι σίγουρο ότι δεν χρειάζεται. Και το δεύτερο που είναι και το κύριο. Η αστική ευθύνη. Εάν αυτά τα FE ρομπότ προκαλέσουν ζημίες. Και εδώ το ψήφισμά μας λέει και καλά και άσχημα. Το καλό είναι υποχρεωτική ασφάλιση και ότι υπόλογο πρέπει να είναι ένα ανθρώπινο άτομο. Αλλά πέρα από αυτό λέει και κάτι άλλο που είναι πολύ πιο ανησυχητικό. Ότι θα πρέπει τα ρομπότ να έχουν ειδική νομική προσωπικότητα. Τώρα αυτά είναι τρομακτικά. Άρα οι άνθρωποι που δημιουργούν τα ρομπότ δεν θα είχαν πλέον καμία ευθύνη. Αυτό είναι αντίθετο σε οποιαδήποτε έννοια ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και βέβαια στο πολύ λογικό ε, ε δικαίωμα των παθόντων να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν αποζημίωση από κάποιο άτομο. Πρόεδρος, ε, έχουμε καθυστερήσει πολύ. Θα συνεχίσουμε ε, για το θέμα αυτό σε κάποια από την επόμενη συνεδριάση μας. Πρόεδρος. Αν είναι να το ξανασυζητήσουμε όταν θα έχουμε περισσότερο χρόνο, καλή ιδέα. Για να συμφωνήσουμε και τι δράση μπορεί να αναλάβει το Κοινοβούλιο. Στην έκθεση ε, βεβαίως ε, απλώς αναφέρουμε τις διάφορες ε, και μάλιστα όλες τις εναλλακτικέ λύσεις. Αλλά όλοι συμφωνούσαμε ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να παραμείνουν εντός του πλαισίου αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Και κάτι ακόμη. Η νομοθεσία μπορεί να επηρεάσει και την τεχνολογία. Το ποιος θα είναι υπόλογος, για παράδειγμα, θα επηρεάσει την εξέλιξη των αυτονόμων οχημάτων. Εάν θα είναι υπεύθυνο ο οδηγός, θα αποφασίζει εκείνος ε, τι πρέπει να περιέχει ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Αν ε, θα είναι υπεύθυνο ο παραγωγός, θα αποφασίζει ο παραγωγός. Να τα ξαναπούμε άλλη φορά. Πρόεδρος, ωραία πρέπει να κλείσουμε τώρα το θέμα αυτό. Θα συνεχίσουμε τώρα τη συνεδρίαση και κλεισμένο των θυρών Οπότε παρακαλώ όσους δεν δικαιούνται να παρακολουθήσουν μια και κλεισμένο το θερών συνεδρίαση να αποχωρήσουν τάχιστα παρακαλώ.